που ε, θα έχουν οι εξελίξεις της σχέσης Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών στις ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Εμείς ε, θέλουμε να υποστηρίζουμε τις δυνατότητες που πρέπει να έχουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στο Ιράν, αλλά ταυτόχρονα παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις έτσι ώστε να ξέρουμε τι θα κάνουμε σε περίπτωση κλιμάκωσης. και επίσης ε, ε, να δούμε τι θα γίνει με την block legislation. Deputy Chief of Staff uh, to the President of the Islamic Έχουμε εδώ έναν εκπρόσωπο της ε, Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ο οποίος είναι και επικεφαλής άλλωστε στην διαπραγματευτική ομάδα του ΣΥΠΙΑΙ. Θα δώσω όμως αμέσως τον λόγο ε, θα του δώσω τον λόγο να εξηγήσει την κατάσταση. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ, έτσι ώστε να ανταλλάξουμε απόψεις για ένα από τα ζητήματα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ε, εξωτερική πολιτική του Ιράν και για την Ευρωπαϊκή Ένωση το κοινό σχέδιο δράσης. Είναι ένα από τα ε, πλέον αυστηρά ε, συστήματα παρακολούθησης επίβλεψης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. 20 εκθέσεις από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας έχουν επιβεβαιώσει ότι το πρόγραμμά μας είναι αποκλειστικά πολιτικής φύσεως. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε πλήρως εκπληρώσει τις ε, δεσμεύσεις μας έναντι του κοινού σχεδίου και περιμένουμε ότι αντιστοίχω θα πρέπει να αποφεληθούμε από αυτό. Δυστυχώ έχουν υπάρξει απόπειρε για να ε, υπονομευθεί αυτή η καλή συνεργασία. Πρώτα απ' όλα με την μονομερή και παράνομη απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να, να αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από το σχέδιο αυτό στην πραγματικότητα αυτό που συνέβη είναι ότι απομονώθηκαν οι Ηνωμένε Πολιτείε και είδατε ότι το Ιράν δεν έκανε το λάθος να βιαστεί. Προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε με, τις με τα υπόλοιπα μέρη, με τη Ρωσία, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους υπολείπους, για να βρεθεί μια λύση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε όχι απλώς αποχώρησαν από αυτή τη συμφωνία, αλλά επίσης ενεργά προσπαθούν να πιέσουν και να πείσουν ακόμα και εκφοβίζοντας άλλα κράτη να τα πιέσουν να μην εφαρμόζουν το διεθνές δίκαιο και να μην εφαρμόσουν την απόφαση 2231 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Προχώρησαν επίσης μόνο μονομερός σε κυρώσεις και απειλούν τα τρί, τις άλλες χώρες ότι θα, τις, θα τους επιβάλλουν κυρώσεις εάν εφαρμόσουν αυτό το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επίσης χρησιμοποιούν την πίεση των οικονομική μέσω του δολαρίου. Η επιβολή αυτών των κυρώσεων είχε ως αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις, ξένες επιχειρήσεις να αποχωρήσουν από το Ιράν. Η επιβολή των κυρώσεων κατά του Ιράν προσπαθεί να δημιουργήσει προβολήματα, δυσκολίες στον πληθυσμό του Ιράν. Αυτό συμπεριλαμβάνει ακόμα και την διατροφική του ασφάλεια. Είναι αδικαιολόγητο αυτό υπό οποιασδήποτε προϋποθέσεις. Είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο και απάνθρωποι πολιτική η οποία θα πρέπει να καταδικαστεί από όλες τις ε, ειρηνικές χώρες. Ε, το, Ιράν τηρεί πλήρως το κοινό αυτό σχέδιο, το οποίο προβλέπει και έχει βασιστεί στην αρχή της αμοιβαιότητας και περιμένουμε τα αντίστοιχα ωφέλη από αυτό. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να αρθούν όλες οι κυρώσεις οι οποίες έχουν επιβληθεί εξαιτία του πυρηνικού προγράμματος και να προχωρήσει η εξομάλυνση των οικονομικών και πολιτικών σχέσεων με το Ιράν. Πρώτο βήμα το που θα πρέπει να έρθει από τις ΗΠΑ να είναι να σταματήσει αυτή, αυτός ο εκφοβισμός, ο παράνομος εκφοβισμός των εταιριών. Επίσης να εφαρμόσουν τη νομικά δεσμευτική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου που ελήφθη στις 3 Οκτωβρίου του 2018. Πιστεύουμε ότι σε αυτή την προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Μέχρι στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι έχει ουσιαστική πολιτική βούληση να εφαρμοστεί το κοινό σχέδιο και να προχωρήσει και να, τη συνεργασία της με το Ιράν επί τη βάση αυτή. Ε, ε, εκτιμούμε τις προσπάθειες που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, θεωρούμε ότι έχει έρθει η ώρα και για πολιτικέ δεσμεύσει και η μετάφραση των πολιτικών δεσμεύσεων σε πραγματικά αποτελέσματα. Οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να σώσουν τη συμφωνία για το πυρονικό μα πρόγραμμα, το οποίο συμπεριλαμβάνει και οικονομικέ πτυχέ, κατά την άποψή μα. Ο μηχανισμό αυτό θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή πριν την καταληκτική ημερομηνία της 4 η Νοεμβρίου. Δεύτερον, θα πρέπει να συνεχιστούν και να προστατευτούν οι επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στο Ιριάν σύμφωνα με το κοινό σχέδιο. Τρίτον, θα πρέπει να επιπεθούν τα ε, ζητήματα της, ε, των εσόδων από την πωλήσει ε, φυσικού αερίου και πετρελαίου από το Ιράν. Μετά θα πρέπει να αναλυφθεί δράση πολιτική ε, στο πλαίσιο του Οργανισμού Ενωμένων από τις ευρωπαϊκές χώρες. Πιστεύουμε ότι η εξομάλυνση αυτών των σχέσεων έχει καθυστερήσει. Θεωρούμε ότι το κοινό σχέδιο είναι μια σημαντική διεθνή κατάκτηση. Το Ιράν έχει τηρήσει όλες του τι υποχρεώσει. Δυστυχώ βλέπουμε ότι άλλα μέρη δεν πράττουν το ίδιο. Το Ιράν έχει λάβει και μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ένα από τα τελευταία ήταν η επικύρωση από το κοινοβούλιο μας της Διεθνούς Σύμβασης για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η παράνομη αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από το κοινό σχέδιο καθιστά την, την θέση των υπολείπων κρατών, των υπολείπων μερών ακόμα πιο σημαντική και ευαίσθητη. Θεωρούμε ότι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και η θέση της είπα της εκπροσώπου ε, ήταν θετική, το αναγνώρισε αυτό και ο εκπρόσωπό μας στη Γενική Συνελευστό ΙΕ, όμως έρχεται η προθεσμία και είναι πολύ σημαντικό εμείς να γνωρίζουμε πώς θα αντισταθμιστούν οι απώλειες από την αποχώρηση που δημιούργησε η αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη στάση που θα επιλέξουν οι Ευρωπαίοι. Ελπίζουμε να καταλήξετε σε ένα λεπτομεριακό και ουσιαστικό σχέδιο έτσι ώστε να σωθεί αυτή η συμφωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω ισπανικά. Βάλτε ακουστικά. Θέλω να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους και θα ήθελα να σας καλωσορίσω από την Επιτροπή Εξωτερικό, γιατί δεν κατάφερα πριν να σας καλωσορίσω. Η Επιτροπή Εξωτερικών, όπως ξέρετε, παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ τις τελευταίες ε, εξελίξεις ό,τι αφορά αυτό το σχέδιο, το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης. Θέλω να εκφράσω εκ νέου την πλήρη υποστήριξη της Ένωσης προς το σχέδιο, γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό στοιχείο της ε, παγκόσμιας αρχιτεκτονικής για τη μη διάδοση. Σημαντικό δε επίτευγμα και για την πολυμερή διπλωματία, το οποίο στηρίζει ομόφωνα το Συμβούλιο ασφαλεία ε, του ΟΗΕ. Με το ψήφισμα 2231 σας καλωσορίζω λοιπόν, σας χαιρετούμε από την Επιτροπή Εξωτερικών και θα σας υποστηρίξουμε, παρακολουθούμε εκ του και δεν θα μακρηγορήσω άλλο, επαναδίνω ξανά το λόγο στον πρώτη της Επιτροπής Εμπορίου. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους βουλευτές. Ένα λεπτό καθένας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις ε, προς προσκεκλημένους. Ας γίνει με μορφή ερώτησης ε, η παρέμβαση του λεπτού. Κυρία Σχάκε, μιλώ εκ μέρους και της Επιτροπής ε, Διεθνών Σχέσεων και της και της Επιτροπής Διεθνού και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο από όλο το πολιτικό φάσμα ότι είμαστε προσιλωμένοι στην πυρηνική συμφωνία και είμαστε απογοητευμένοι που αποχώρησε η Αμερική από την παγκόσμια κοινότητα. Το θέμα είναι να μπορούν να γίνονται οι επιλογές. Μέγιστη ελευθερία της επιλογές που, πρέπει να είναι και προτεραιότητα μας. Μόνο τους θα πρέπει να δουν ε, πώς ε, θα ε, προχωρήσουν μέσα στη νέα πραγματικότητα. Υπάρχουν επιχειρήσεις που θέλουν και άλλες που δεν θέλουν να κάνουν να έχουν δραστηριότητα στο Ιράν. Το θέμα είναι ότι η Αμερικανική αποχώρηση πρέπει να αντισταθμιστεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως παραμένει δεσμευμένη, προσιλωμένη, έχει ξεπεράσει, για να μην πω έχει πάρα ξεπεράσει τα όρια για να αντισταθμίσει ε, την αποχώρηση των πακέτης κυρώσεων. Δεν μπορούμε λοιπόν να πιέζουμε περισσότερο, είναι κάτι απαράδεκτο, δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό, ότι εμεί πρέπει να κάνουμε παραπάνω. Και ένα τελευταίο σχόλιο, απαντώντα ε, σε αυτά που είπατε για τα προβλήματα και τι δυσκολίε ε, που έχετε να αντιμετωπίσει ο ιρανικό πληθυσμό με τι νέε Αμερικανικέ κυρώσει φυσικά και θα πρέπει αυτό να το αποφύγουμε. Στρέφομαι όμως στους ηγέτες Ισλαμικής δημοκρατία. Αυτοί είναι οι πρώτοι που πρέπει να ξεκινήσουν να σέβονται τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Και αυτό θα βοηθήσει πολύ περισσότερο από ότι ε, κακό κάνουν οι αμερικανικές κυρώσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει η κυρία Ζαήφη. Ήθελα να πω ότι οι κυρώσεις του Προέδρου Τραμπ είναι μονάχα ένα από τα σκέλη της πολιτικής του που βασίζεται στην ε, διαρκή πίεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αρκεστεί σε μια αμυντική ε, στάση. Αν θέλει πραγματικά να ε, κερδίσει αξιοπιστία απέναντι στους εταίρους, θα πρέπει να έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ισχυρή θέση και να πάρει μέτρα κατά Αμερικών, αμερικανικών επιχειρήσεων. Πέρα από την χρήση της δυνατότητας εμπλοκής μπορεί να εισαγάγει και νέα μέτρα. Η χρήση του ευρώ για τις διεθνείς συναλλαγές φαίνεται κάτι προφανές και θα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχύσει τη θέση του ε, στην διεθνή χρηματοπιστωτική αγορά. Προς τα εκεί θα πρέπει να κινηθούμε. Τέλος, όσον αφορά ε, το πεδίο εφαρμογής ε, του νόμου εμπλοκής, θα πρέπει οπωσδήποτε να διευρυνθεί. Αναφέρομαι κυρίως σε αντίστοιχες αμερικανικές διαδικασίες οι οποίες υποχρεώνουν τις Αμερικανικές αμερικανικές επιχειρήσεις να αποκαλύψουν στην κυβέρνηση ε, λεπτομέρειες ε, των εμπορικών τους ε, συμφωνιών έναντι κυρώσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής. Πρώτον, όλες οι διεθνείς ε, οργανώσεις, ε, λέει ο κύριος Νάρτ, ε, πρέπει να εφαρμόσουν τη συμφωνία. Δεύτερον, είναι προφανές ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ακολούθησαν την πεπατημένη Τραμπ, που δεν είναι America First, αλλά America Alone. Νομίζω ότι αν θέλουμε να είμαστε αξιοπρεπείς, θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιδράσουμε η στρατηγική της Βόρειας Αμερικής ε, είναι ε, αντιπαράθεση και με το Ιράν και με άλλες γειτονικές χώρες, είναι προφανές αυτό. Επομένως εδώ δεν ε, συζητούμε εάν οι Ηνωμένε Πολιτείε θεωρούν ότι το Ιράν καλύπτει ή όχι τις υποχρεώσεις. Εν πάση περιπτώσει, εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουμε όχι φιλοσοφικές τοποθετήσεις, αλλά συγκεκριμένες απτές και τοποθετήσεις και να αντιδράσουμε αντιδράσουμε σε αυτό που είναι προφανές ότι είναι ε, ε, ε, αμερικανική, αμερικανικός εκβιασμός βάσει αυτής της νέας πολιτικής Τραμπ που βλέπει τον εαυτό του σαν παγκόσμιο αυτοκράτορα εάν εμείς δεν έχουμε την δυνατότητα όχι να ε, πιέσουμε βάσει των ε, οικονομικών προβλημάτων που μπορεί να έχουν επιχειρήσεις, αλλά δεν είμαστε, λέω, σε θέση εμείς να δημιουργήσουμε πολιτική γραμμή, τότε τι να σας πω. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει η κυρία Φορέντζα συμφωνούμε με την θέση της ε, Φεντερίκας Μογκερίνη στα Ηνωμένα Έθνη τον ε, Σεπτέμβριο, δηλαδή δημιουργία, ενεργοποίηση ενός επιπλέον οικονομικού μηχανισμού ε, για να βοηθηθεί το Ιράν, το οποίο έχει πληγεί από τις αμερικανικές κυρώσεις. Η απόφαση του Προέδρου Τραμπ να αποσυρθεί από την συμφωνία με το Ιράν αποτελεί ε, κίνδυνο για ολόκληρο τον κόσμο. Ευελπιστούμε ότι αυτό το νέο εργαλείο δεν θα χρησιμοποιηθεί μονάχα για το Ιράν, αλλά και για όλες ε, τις χώρες οι οποίες υφίστανται εξωχωρικές ε, πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ας πούμε η Κούβα. Πολλές είναι οι επιχειρήσεις οι ευρωπαϊκές οι οποίες φοβούμενες ε, τα ε, αντίπεινα της, Ευρω... Αμερικής θέλουν να αποσυρθούν από το Ιράν. Δεν είναι δυνατόν να ακολουθήσουμε αυτήν την εμπορική βουλημία του Προέδρου Τραμπ. Δεν είναι δυνατόν να τον ακολουθήσουμε στις ε, πιέσεις του. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει απλώς να βοηθήσουμε τις δικές μας ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιχειρήσεις, αλλά θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις ε, του ε, Προέδρου Τραμπ. Διαφορετικά θα πρέπει και εμείς να κάνουμε τα ίδια, αντίπεινα δηλαδή στις αμερικανικές ε, επιχειρήσεις οι οποίες δρούν στην Ευρώπη. Οι Mr. Mr. ευχαριστώ. Α είμαστε ξεκάθαροι πρώτα απ' όλα. Δεν πρόκειται μόνο για τι ΗΠΑ. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει εμπλοκή. Μάλλον είναι ξεκάθαρο, μα λένε οι Ισραηλινέ μυστικέ υπηρεσίε, ξεκάθαρα ότι το Ιράν παραβιάζει τη συμφωνία συστηματικά. Ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ τη συνάδελφο που αναφέρει το απαράδεκτο, την απαράδεκτη κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν. Ανησυχούν για άλλε χώρε οι συνάδελφοι, γιατί δεν ανησυχούμε εξίσου και για το Ιράν. Τρίτον, το Ιράν συστηματικά έχει αποστεθερεοποιήσει ή έχει επιδιώξει να απαστεθερεοποιήσει την περιοχή της Μέσης Ανατολής και εμπλέκεται στην κατάσταση στη Συρία. Παρά το γεγονό μάλλον εξαιτία του γεγονότος ότι έχουμε αυτή την απέχθεια προς τον πρόεδρο Τραμπ, δεν βλέπουμε καθαρά. Δε, αυτή η αλαζονία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, των υπηρεσιών της, έχει ως, είχε ως αποτέλεσμα να διχαστεί η Δύση. Και οι Ιρανοί δεν πιστεύουν στην τύχη τους. Γι' αυτό μη Thank you for our uh, Iranian friends for coming here. I have two very short questions. Έχω δύο απλές ερωτήσεις, γνωρίζοντας ότι η ομάδα των σοσιαλιστών ήταν από εκείνες τις πολιτικές ομάδες που συστηματικά υποστήριξαν την Συμφωνία για το Πολιτικό Πρόγραμμα του Ιράν. Το πρώτο μου ερώτημα είναι, ποια είναι η δικιά σας αξιολόγηση όσον αφορά την σταθερότητα στην περιοχή και δεύτερον, τι, πώς προβλέπετε να εξελιχθούν οι σχέσεις σας με την Σουηδική Αραβία και το Ισραήλ, τώρα πια που βλέπουμε ότι και οι Ηνωμένε Πολιτείε προσεγγίζουν τη σχέση του με τη Σουαουδική Αραβία με βάση την προαιώνια σύγκρουση μεταξύ Σουνιτών και Σιητών. Ευχαριστούμε. Εγώ θα μιλήσω προσωπικά χωρίς να μην εκπροσωπώ την ομάδα μου. Πάντοτε υποστήριζα το κοινό πλήρες σχέδιο ως το μόνο τρόπο για να περιορίσουμε τους ε, κινδύνους ενός πυρηνικού προγράμματος ε, εκτός ε, διεθνούς ε, ελέγχου από το Ιράν. Συμφωνώ με τον συνάδελφο ότι το Ιράν έχει απαράδεκτη κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως και άλλες χώρες στην περιοχή, όπως για παράδειγμα η Σαουδική Αραβία. Πρόσφατα είχαμε αυτή την αξαφάνιση, πιθανότατα απαγωγή ενός Σαουδάραβα δημοσιογράφου που είχε επισκεφθεί το προξενείο της χώρας στην Κωνσταντινούπολη. Επομένως, εγώ το βλέπω το ζήτημα διαφορετικά. Προσπαθούμε να, να έχουμε περιορισμό τη διάδοση των πυρηνικών όπλων και ιδιαίτερα μια σύγκρουση με πυρηνικά όπλα στη Μέση Ανατολή, κάτι που θα ήταν ε, τραγική. Δεν έχω δει εγώ αποδείξεις ότι παραβιάζει το Ιράν τις προβλέψεις του ε, κοινού σχεδίου έχουμε κάποια στοιχεία για βαλιστικούς πυράβλους, αλλά όχι για τις προβλέψεις του σχεδίου. Ίσως αυτές να πρέπει να ενισχυθούν. Πιστεύω λοιπόν ότι η στάση των ΗΠΑ είναι καταστροφική και πιστεύω ότι αυτό ε, εντάσσεται και σε ένα γενικότερο πλαίσιο που προσπαθεί να βάλει το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit να πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στο εάν θα συμμετάσχει σε αυτό το νέο κλαμπ που φαίνεται διαμορφώνεται με τον Καναδά, με τις ΗΠΑ ή θα να έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα θα λάβω το λόγο ως εκπρόσωπος της Γκουε και της Ενωμένης Αριστεράς και όχι ως αντιπρόεδρος της ΑΦΕΤ. Συγχαρητήρια καταρχάς πρώτη κοινή δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, για μια, μετά από μια συνθήκη για τη μη διάδοση και υπέρ της σταθεροποίησης μιας περιοχής που αποσταθεροποιήσαμε δυστυχώς πολλές φορές εμείς οι Ευρωπαίοι και είναι σαφές ότι δεν είναι η πρώτη φορά που είπα απειλούν ε, τράπεζες και επιχειρήσεις από την Ευρώπη. Το είδαμε και με το εμπάργκο στην Κούβα. Για πρώτη φορά όμως βλέπω οι περισσότερες ομάδες ε, να ε, σκέφτονται να ανταποκριθούν σε περίπτωση και να αντιδράσουν σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα με ε, ευρωπαϊκή εταιρεία που δραστηριοποιείται στερα. Πολλές φορές ο Τραμπ ή η Σαουδική Αραβία μιλά για το σχέδιο βαλιστικών πυράβλων, το χρησιμοποιεί ως πρόσχημα. θεωρητικά υποτίθεται ότι απειλεί μέχρι και την Ευρώπη. Επτά μυστικέ υπηρεσίε. λένε ότι κανένα από του βαλιστικού όμω πυράβλου αυτού, δεν έχει τέτοιο βελικές που να μπορούσε να φτάσει στην Ευρώπη. Έχετε κάτι να μα απαντήσετε. Πρόεδρο, ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο στον προσκεκλημένο μας ε, για να απαντήσει σύντομα. Ε, δύο λεπτά μόνο έχετε αν θέλετε, για να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις. Thank you. Thank you very much, Mr. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές για τα σχόλιά τους. Ακόμη και αυτούς που δεν, τους, ε, δεν συμφωνώ με αυτά που είπαν. Επειδή δεν έχω χρόνο, θα ήθελα να δώσω στις απαντήσεις στα διάφορα θέματα που ήγηραν οι βουλευτές. Σε ό,τι αφορά τις που θα αντιμετωπίσει ο ελληνικός λαός. Αυτό που θέλω να πω ήταν ότι οι κυρώσεις έχουν ακριβώς σχεδιαστεί από του Αμερικανούς έτσι ώστε να προκαλέσουν δυσκολίες ε, στον Ιρανικό λαό. Και επομένω, χρέος οποιοδήποτε ανθρώπου στον πλανήτη γη είναι να αντιταχθεί στο Αμερικανικό αυτό σχέδιο γιατί στόχο έχει να πλήξει τους ε, ε, άμαχους. Ποιος είναι αυτό ο οποίο θα πληγεί λόγω έλλειψη φαρμακών και τροφίμων γιατί λένε ότι αυτά εξαιρούνται. Όταν όμως ε, δημιούργησαν τα προβλήματα με τις τράπεζες, τις δικές μας επιχειρήσεις που δεν μπορούσαν να έχουν συναλλαγές με άλλες εταιρείε και με ευρωπαϊκές κτλ. Λένε ότι δεν θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα στον απλό λαό. Μιλάμε όμως για ένα πραγματικό, απτό πρόβλημα. Κάτι άλλο ήταν η χρήση του ευρώ for European Όπως είπα, είπα, προσπαθούν να χρησιμοποιούν το δολάριο ως ε, πυρομαχικό. Άρα εμείς προσπαθούμε να ε, ε, παρακάμψουμε αυτό το πρόβλημα για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με ευρωπαϊκές και τα λοιπά. Αυτοί χρησιμοποιούν ως όπλο το νόμισμά τους και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ένα άλλο σημείο ήταν κατά πόσον σέβεται και τηρεί τη συμφωνία το Ιράν και είναι πραγματικά ε, παράλογο να ακούγεται ότι δεν τη σεβόμαστε αυτή τη συμφωνία γιατί ο Κρητής είναι η εταιρεία η Διεθνής ε, Οργάνωση Ατομικής Ενέργειας η οποία λέει ε, ακριβώς ποιος τηρεί και ποιος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του. Συμφωνώ λοιπόν, με, μάλλον δεν συμφωνώ με τον ισχυρισμό ότι εμείς παραβιάζουμε το σχέδιο. Σε ό,τι αφορά τους πυράβλους. Δεν υπάρχει διεθνή συνθήκη για τον περιορισμό της χρήσης πυράβλων. Το Ιράν έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Άλλοι χρησιμοποιούν τα χρήματά τους, δισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται. Δείτε τι γίνεται στην Ιεμένη, δίπλα μας, στη γειτονιά μας. Ποιος στέλνει όπλα στη Σαουδική Αραβία που χρησιμοποιούνται κατά αμάχων, κατά αθώου πληθυσμού και στην Ιεμένη και αλλού. Εμείς χρησιμοποιούμε τις δικές μας εγχώριες ικανότητες και δυνατότητες για αυτοάμυνα. Άλλες γειτονικέ χώρες ε, με τη βοήθεια των φίλων της από την Ευρώπη και τη ΣΥΠΑ δημιουργούν πολλά προβλήματα στην ε, γειτονική περιοχή. Άρα, κατά την άποψή μας έχουμε και εμείς κάθε δικαίωμα να υπερασπιστούμε αυτούς Σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ουδής τέλειο. Δείτε τι γίνεται γύρω σας, παντού. Αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι κάθε ευκαιρία που μας δίνεται να την αξιοποιήσουμε για να βαθμίζουμε, να διατηρούμε και να σεβόμαστε τις δεσμεύσεις μας, αλλά ως μουσουλμάνοι έχουμε το δικαίωμα να προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και κάνουμε πάντα το δυνατόν προς αυτήν την κατεύθυνση. Όσοι ρωτάνε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μήπως εθελοτυφλούν και κλείνουν τα μάτια τους απέναντι στην έλλειψη φαρμάκων και τροφίμων, που ακριβώς στόχο έχει να δημιουργήσει πιέσει στον Ιρανικό λαό. Είναι λίγο παράλογο, αλλά αυτά ευχαριστώ, Πρόεδρο. Σα ευχαριστώ και κύριο Περμούη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστήσω όλε και όλου όσοι συμμετείχαν σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση καλή επάνωδο στην Τεχεράνη για την αρνητική αντιπροσωπεία, ένα θέμα που θα συνεχίσει να μας απασχολεί στη συνέχεια. Ευχαριστώ, ολοκληρώσαμε. Indeed, and Ωραία. Θα διακόψουμε για ένα λεπτό, λέει ο Πρόεδρος, γιατί θα περάσουμε μετά στο σημείο 9, που είναι η, η συνάντηση των συντονιστών, συνεδρίαση των συντονιστών, συγγνώμη, ε, επίσης για κλεισμένο των θυρών.